αύριο. Επίσης σας λέγω ότι το ΕΛΚ έχει υποβάλει τα ε, ακόλουθα αιτήματα. Ο κύριος Αντώνιο Καντσάν, μέλος της Αντιπροσωπείας για σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο, θα αντικαταστήσει ο κύριος Αλφρέντο Αντωνιώτσι. Ο κύριος Αλφρέντο Αντωνιώτσι ε, θα, αντιπροσ... θα αντικαταστήσει ο κύριο Καντσάν στην ε, κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Κροατίας. Επίσης, ο κύριος Ανδρέα Κατσολίνα θα γίνει μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών μετά από αίτημα των Σοσιαλιστών. Κύριε έχετε κάποιο πρόβλημα. Όχι, όχι. Κανείς λοιπόν δεν αντίθεται στις προτάσεις ε, αυτές. Τα πρακτικά της ε, παρούσας συνεδρίασης ε, θα υποβληθούν στην έκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επόμενη συνεδρίαση. Αν δεν έχει κανείς αντίρρηση, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών τη σήμερα θα μεταδοθούν ως ήθιστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ εις το μόνο σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.